εργασιών για αυτή την εβδομάδα. Από την διάσκεψη των Προέδρων, αμέσως κύριε Πόσελ, θα σας δώσω τον λόγο αμέσως. Σύμφωνα με το άρθρο 137 του κανονισμού, στις 7 Μαρτίου εγκρίθηκε το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης και το οποίο έχει διανεμηθεί. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιες προτάσεις για τροποποίηση αυτού του σχεδίου εργασιών ημερήσιας διάταξης. Κύριε Πόσελ, έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Με μικρόφωνο τώρα κύριε Πόσερτ. Στην Επιτροπή Εξωτερικών εδώ και μήνες έχουμε σημαντικές εκθέσεις που προετοιμάσαμε για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα θέματα και της Σερβίας και του Κωσυφοπεδίου. Αυτές οι εκθέσεις εδώ και μήνες είχαν προβλεφθεί για την Τετάρτη το απόγευμα, το βράδυ. Έχουμε και αντιπροσωπείς κυβερνήσεων και κοινοβουλίων, ειδικού δημοσιογράφους και διπλωμάτες που έχουν προσέθει στο Στρασβούργο ειδικά για αυτό το θέμα. <clears throat> Τώρα, την Πέμπτη το απόγευμα, χωρί να το γνωρίζουν οι κοινοβουλευτικέ ομάδε, από τη διάσκεψη των Προέδρων αυτό το θέμα αποσύρθηκε από την ημερησία διάταξη. Σύμφωνα με το σύστημα του Ανατολίτικου Παζαριού. Κάθε πρόεδρο κοινοβουλευτική ομάδα είχε κάποια πρόταση και είπαν ότι από την Αίγυπτο στην Ουκρανία θα υπάρξουν ε, αλλαγέ και θα ενταχθούν όλα αυτά τα θέματα για την περίοδο συνόδου του Απριλίου. Θέλω να διαμαρτυρηθώ για αυτό το γεγονό και θέλω να απευθύνω έκκληση στην διάσκεψη των Προέδρων να εργάζονται με σοβαρότερο τρόπο μελλοντικά και να μην ακολουθούν τέτοιες διεργασίες. Κύριε Πόσερτ, ως ε, πολιετές μέλος της διάσκεψης των Προέδρων, πρέπει να σας πω να μην <laughs> προσβάλλετε το περσικό ανατολίτικο παζάρι με τέτοιο τρόπο, με τέτοιες συγκρίσεις. Υπήρξε πληθώρα, πρέπει να πω, πολυάριθμοι σοβαροί λόγοι που οδήγησαν σε αλλαγή της ημερήσιας διάταξης εργασιών. Δεν επιθυμώ και ούτε μπορώ να ε, ε, διευκρινίσω όλους αυτούς τους λόγους. Για αυτούς όλους τους λόγους ε, αναβλήθηκαν για την επόμενη περίοδο συνόδου αυτά τα θέματα. Όμως σημειώνουμε τη διαμαρτυρία σας. Για τη σημερινή ημερήσια διάταξη της Δευτέρας υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις ή προτάσεις. Παρακαλώ εσείς. Θα ήθελα να προτείνω η συζήτηση για την ένταξη τη Σερβίας και του Κωσυφοπεδίου να καθιστά όχι για τον Απρίλιο του 2013 αλλά για τον Απρίλιο του 3000. Αγαπητέ συνάδελφε, κύριε συνάδελφε, η χρονική διάσταση του αιτήματό σα είναι σχετικά μεγάλη και γενναιόδορη. Θα έπρεπε να είχατε θέση μέχρι τι 4 το αίτημά σα. Κατά τούτο και οι δύο αυτέ ε, χρονικέ διαστάσει ε, δεν είναι οι διαδομένε, οι πιο εύθετε. Λοιπόν, υπάρχουν άλλοι. Ο κύριο Οντί, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρετε, παίρνω πολλές φορές το λόγο το θέμα αυτό, γι' αυτό και δίσταζα. Την Δετάρτη θα μιλήσουμε για το επόμενο Συμβούλιο και την ίδια ώρα θα μιλήσουμε και για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Έχουμε καλέσει τον πρόεδρο Βαν Ρομπόη. Εάν ναι, γιατί δεν θα είναι παρόν, αρνείται να έρθει. Θεωρώ ότι η Τετάρτη το πρωί θα ήταν πολύ σωστή στιγμή παρουσία του Πρόεδρου Βαρομπόη να συζητήσουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου και να ακούσουμε και την άποψή του για το Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας. Λυπούμε λοιπόν που δεν θα είναι παρόν ε, ο Πρόεδρος και θα ήθελα να ξέρω αν ε, εμείς δεν επιμείναμε ή αν εκείνος αρνείται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Οντή. Ξέρετε κύριε Οντή ότι υπήρξε μια έκτακτη ανοιχτή συνεδρίαση των Προέδρων όπου ο κύριος Φαν Ρόμποϊ αμέσως μετά τη Σύνοδο Συμβουλίου άμεσα εξέθεσε αυτά τα συμπεράσματα και αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν η συζήτηση την Τετάτη θα είχε δώσει κάποια περισσότερα αποτελέσματα από τα όσα εξετέθησαν κατά αυτή την έκτακτη συνεδρίαση. Κατά άλλα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου την ε, Τετάρτη. Έχουμε επίσης και, την, το Συμβούλιο της Πέμπτης που προετοιμάζεται από πλευράς του. Και πάλι θα συζητήσω αυτό το θέμα με τον κύριο Φαν Ξέρουμε με τι ε, ζήλο αγωνίζεστε για να προσέλθει εδώ. Όμως κύριο Ντί είσαστε μόνος σας σε αυτόν τον αγώνα που δίνετε πρέπει να σας πω. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να παρέμβουν για την ημερήσια διάταξη. Όχι, εντάξει. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη εργασιών μας για σήμερα. Και ξεκινάμε τώρα με την κοινή συζήτηση για την Διεθνή ημέρα της γυναίκας. Παρακαλώ κύριε Κένρικαν, έχετε τον λόγο. Το μικρόφωνο, πρέπει να πάρετε ένα μικρόφωνο. Uh, uh, uh, Ήθελα να πω ότι εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο γίνεται μια διάκριση κατά της εθνικής γλώσσας της δικής μου χώρας των Ιρλανδικών γίνεται εδώ και έξι χρόνια. Έχει μια ιστοσελίδα το κοινοβούλιο σε 22 χώρες και υπάρχει μία γλώσσα που είναι απούσα από αυτό το νηστότοπο. Είναι διαθέσιμη στο Συμβούλιο Υπουργών και στην Κομισιόν παρόλα αυτά. Μάλιστα, εντάξει. Κύριε Γκάλαγκερ, όμω αυτό σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή την ολομέλεια, σε αυτή τη συζήτηση δεν μπορεί να α, αναφερθεί κανεί για ένα θέμα το οποίο δεν εγγράφεται στην ημέρησια διάταξη και δεν τίθεται υπό συζήτηση Κατά τα άλλα, είσαστε σε επαφή μαζί μου για τον ιστότοπο αυτό. Δεν έχει εγγραφεί στην ημερησία διάταξη. Μπορείτε να συζητήσετε ευχαρίστω διμερό μαζί μου αυτό το θέμα αυτού του ιστοτόπου. Θα σα εισακούσουν, θα εισακουστείτε και θα ληφθεί υπόψη αυτό το έτοιμά σα, αλλά συζητούμε τώρα για τη διεθνή ημέρα γυναικών. Θα λάβει τον λόγο ως εισηγήτρια η κυρία Μωράν Σαρτιέ. Παρακαλώ κυρία Μωράν Σαρτιέ. Πού είναι η κυρία Μωράν Σαρτιέ. Παρακαλώ κυρία, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να χαιρετήσω την Βιβιάν ε, Ρέντινγκ, αντιπρόεδρο της ε, Επιτροπής, η οποία Επίσης.